βρισκόμαστε πάνω κάτω στο προβλεπόμενο ωράριο, θα φροντίσουμε να σεβαστούμε τι χρονικές προθεσμίε. Έχουμε μεσά μα τον στρατηγό Μωρή Τεντεζό, πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα του δώσω το λόγο ολίγου. Θα ήθελα να σα πω πω τα πρακτικά των συνεδριάσεων 20 και 21 Ιουλίου έχουμε τη διάθεσή μα και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει μας το τέλο τη συνεδριάσεω, θα θεωρηθούν ω συγκεκριμένα. Επίση να παρατηρήσω πως στις ε, προ... επόμενη συνεδρίασή μας στις 15.00 θα υποδεχθούμε τον ε, Σουηδό πρέσβη, πρόεδρο της ΚΟΠΣ, ε, αλλά και την κυρία Τζανέλα που είναι ε, Πρόσωπο ε, για την, στην Επιτροπή για την καταστροφή ομβλομαζικής ε, καταστροφής, τον κύριο Χάβερ επικεφαλής του ΣΕΠΕΣΕΣΕ, στο πλαίσιο των συναντήσεων που οργανώνουμε με την γραμματεία του Συμβουλίου για να έχουμε ενώπιον της Επιτροπής μας πολλούς επικεφαλής αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχω κατά νου ιδιαίτερα την αποστολή στο Κωσυφοπέδιο. Θα δεχτούμε τον στρατηγό Μερών Και τον Οκτώβριο τον κύριο Μερόκ για την Σάβρεση και αυτός ενώπιον της Επιτροπής μας. Η συνεδρίασή μας ε, εκπέμπεται μέσω web stream, μέσω διαδικτύου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τώρα κάποιους περιορισμούς που έχουμε από γλωσσικής πλευράς, τα δανέζικα, τα λετωνικά, τα σλοβακικά, τα δανέζικα και τα εστονικά δεν ε, τα έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας σε επίπεδο διερμηνίας. Επενθυμίζω ότι χρησιμοποιούνται στη Γερμανία μόνο οι γλώσσε των τακτικών μελών. Μετά από τον κύριο Μπετενζά θα υποδεχτούμε τον κύριο ε, Ιουρέκ. δυστυχώ ο κύριος Μπελουάρ δεν θα μπορέσει να έρθει διότι έχει κάποιες άλλες ε, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Έχουμε ανάμεσα μας τον στρατηγό Μπέτεν Ζακ, ε, που πρόεδρο της Θεωρητικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, επιτροπή αυτή που στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προτού να προωθήσει τις διάφορες στρατιωτικές δραστηριότητε. Ο στρατηγός Μπέτεν Ζακ, που όλοι γνωρίζετε, είναι άτομο το οποίο εκτιμάμε ιδιαίτερα. Έχει εποπτεύσει τις δραστηριότητες μας και τις επιχειρήσεις στο Τσάντ αλλά και στην επιχείρηση Αταλάντη αλλά και την ε, τα δραστηριότητες μας στην ε, Βοσνία. Ο στρατηγός Μπετενζάτ ε, θα αποχωρήσει τον Νοέμβριο, θα αντικαθιστεί από τον Σουηδό στρατηγό Σιρένα και θεωρήσαμε πως θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εμπειρίες του και να προσφέρουμε στον κύριο Πεντεζάτη την δυνατότητα να ανταλλάξει μαζί μας απόψεις ε, σχετικά με την ε, ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και ο κύριος Μπεντεζάρ θα μπορούσε να μας μιλήσει για το μέλλον της ΠΕΣΤ εκτός από τον ε, απολογισμό των 10 ε, ετών της ΕΠΑ. Παρακαλώ κύριε Στρατηγή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που με προσκαλέσατε να παρουσιάσω στην υποεπιτροπή σας την στρατιωτική πτυχή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Για μένα αποτελούσε ανέκαθεν προνόμιο και τιμή να ανταλλάσσω απόψεις με τα μέλη της υποεπιτροπής σας προσφάτως και με ιδιαίτερο διακριτικό τρόπο ε, γιορτάσαμε τα 10 χρόνια από την Συμφωνία της Κολονίας που μας οδήγησε στην διαχείριση των κρίσεων οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλειά μας ε, λαμβάνοντας φυσικά και εφαρμόζοντας τις αρχές οποίες πιστεύουμε. Ε, προωθήσαμε κάποιες στρατιωτικέ δραστηριότητε, βελτιώσαμε τις ικανότητές μας και θα ήθελα να ε, αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, η ΕΠΑ είναι πολύ πιο νέα από ό,τι μπορούμε να πιστεύουμε. Το έτος ίδρυσης είναι στην ουσία το 2003. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια, ε, πρώτε ανθρωπιστικέ δράσει στην Βοσνία και στρατιωτικέ στα Βαλκάνια και στην Αφρική. Λοιπόν, σε έξι χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει έξι στρατιωτικές δραστηριότητες και δεκάξι δραστηριότητες πολιτικής φύσεως. Ένας απολογισμός πράγματι εντυπωσιακό, μοναδικός θα λέγαμε, διότι αυτές οι δράσεις αποτέλεσαν στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυχία, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ε, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, εξάλλου προσφέρει μια προσθέμενη αξία στην διεθνή κοινότητα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί με το ΝΑΤΟ, δεν έχει εξάλλου ούτε τους στόχους ούτε και τα στρατιωτικά μέσα του ΝΑΤΟ. Αλλά η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ισχυρή για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για την πρώτη και μοναδική οργάνωση που μπορεί να προσεγγίσει συνολικά και να διαχειριστεί τις ε, κρίσεις. Π.χ. η Βοσνία Ζεγοβίνη το 2004 οι δραστηριότητε ε, των στρατιωτικών δυνάμεων και των αστυνομικών δυνάμεων συντονίζεται συνεχώς από τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο παράδειγμα, η δράση U4 στο Τσάντ και στην Κεντρική Αφρική στο σύνολό της ε, σχεδιάστηκε από την Γενική Γραμματεία, την Κομισιόν και έτυχε διαχείρισης ε, επιτόπου ε, από τον ειδικό εκπρόσωπο. Η, δράση, ε, η επιχείρηση Αταλάντη οφείλει την επιτυχία της σε μια απόλυτα συντονισμένη δράση αυτή εξ αρχής ανάμεσα στην Κομισιόν για την Γραμματεία του Συμβουλίου και την, το Αρχηγείο. Αλλά ένας άλλος λόγος της επιτυχίας οφείλεται στο ότι σε πολλές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μοναδικός ε, παίκτη ε, διεθνώς αποδεκτός και αυτό έγινε και στην περίπτωση του Τσάντ. Τώρα για να επανέλθω στις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεκινώντας από την Βοσνία της Εγωβίνη, η U4 ε, ξεκίνησε το 2004 για να συνεχίσει μια δραστηριότητα του ΝΑΤΟ που στηρίζεται στα μέσα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη συμφωνία του Βερολίνου, ΣΥΝ, και συμμετέχουν σε αυτήν 2.200 ε, άνδρες. Η κατάσταση είναι ήρεμη, δεν βλέπετε καν μια επικίνδυνη δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον, γι' αυτό λοιπόν προβλέπουμε να μετεθέσουμε αυτήν την δύναμη σε μια δύναμη υποστήριξη ε, ε, των βοσνιακών στρατιωτικών δυνάμεων. Ξέρετε όμως η κατάσταση στην Βοσνία αυτή την περίπτωση έχει λίγο ε, εγκλωβιστεί και πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες ε, σημαντικές εξελίξεις. Θα εξετάσουμε το θέμα του διορισμού ενός ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει ενδεχόμενα διευρυμένες ε, αρμοδιότητες. Η απόφαση αυτή δεν νομίζω θα μπορέσει να ληφθεί τον Νοέμβριο όπως προβλέπετε, διότι τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχει γίνει καμία πρόοδος αφορά το θέμα της ε, μεταφοράς ε, κάποιων θησιδίων αλλά και το καθεστώς του Μπερσκό. Τώρα, αν ε, δεν ληφθεί η απόφαση για το κλείσιμο του γραφείου, Τώρα θα είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να, τροποποιήσει την U4 σε μια συμβουλευτική επιτροπή, διότι θεωρούν ότι ο, ο ύπαρος θα πρέπει να την χάνει τη στήριξη των στρατιωτικών δυνάμεων. Λοιπόν, ορισμένε χώρες που συνεισφέρουν και που έχουν κουραστεί να προσφέρουν στρατιωτικές δυνάμεις από το 1995 άφησαν να εννοηθεί ότι θα αποσύρουν τη συμμετοχή τους εν πάση περιπτώσει το, στα τέλη του έτους. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύριος Σολάνα προσφάτως ε, τόνισε τον κίνδυνο που θα παρουσίαζε η μονοπλευρή απόσυρση για θέματα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας ε, της επιχείρησης. Τώρα, Αταλάντη. Αυτή η επιχείρηση κατά της πειρατείας ε, ανοιχτά της Σομαλίας ξεκίνησε το 2008. Ε, διοικείται από τον ε, στρατηγό, τον ε, Ναύαρχο Χάρτσον και τώρα συμμετέχουν 11 φρεγάτες, κορβέτες, τρεις ε, περιπολίες ε, ναυτικές, ένα αεροπλάνο AWACS, ε, αλλά δυστυχώς δεν διαθέτουν πλοία ανεφοδιασμού. Δεν είναι η μοναδική δύναμη που δράσει στην κόλπο του Άντεν. Υπάρχει και η CTF 151 που διοικούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ, αλλά και φρεγάτες κινέζικες, ινδικές, Σαουδική Αραβία, Ρωσία κλπ. Πάνω από 30 πολεμικά σκάφη λοιπόν βρίσκονται στην περιοχή. Ο συντονισμό ασφαλίζεται μια ομάδα επαφή που βρίσκεται υπό την αιγίδα των ΟΗΕ και στη θάλασσα υπάρχει ένας μηχανισμός άτυπος, το ΣΕΛ, που διαδίδει τις προφορίες σε, όλες σε όλα τα σκάφη και αποφεύγουν οι επικαλύψεις. 217.000 τόνοι ε, τροφίμων έχουν χορηγηθεί στην ε, Σομαλία από τα σκάφη ΠΑΜ που συνοδεύονται από τι δυνάμεις της ε, Αταλάντης. Οι ναυτικές μας δυνάμεις έχουν συνοδεύσει 40 σκάφη, τα υπόλοιπα τα έχουν συνοδεύσει τα σκάφη του ΝΑΤΟ. Εξάλλου εξασφαλίζαμε την προστασία έξι ε, πλοίων ανεφοδιασμού. Τώρα, σε ό,τι φορά τις επιθέσεις, 111 προσπάθειες ε, ε, έγιναν και 48 είχαν, είχαν αισιοπέρας και αλλά το 2009 η επιτυχία αυτών των ε, επιθέσεων των πειρατών μειώθηκε σε 28. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει περιοριστεί σημαντικά με επιτυχία τους ε, βρίσκεται κάτω του 25%. 68 πειρατές έχουν συλληφθεί από την UNAFOR και έχουν μεταφερθεί στην Κένια προκειμένου να δικαστούν η UNEFOR, ε, η Αταλάντη, αν θέλετε, είναι αναγνωρισμένη από τις διεθνείς οργανώσεις και από τους ε, εφοπλιστές ότι είναι η πιο αποτελεσματική δύναμη που έχει δράσει στην περιοχή. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο σαφές και πλήρες ε, σε ό,τι φορά την εμπλοκή τους και υπάρχουν συμφωνίες με όλες τις παράκτες χώρες, με συμφωνία με την Γένεια για την ε, μεταφορά και την ε, δίκη των πειρατών, συμφωνίες ε, με διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς αλλά και με εφοπλιστές. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο, δηλαδή να βρίσκουμε πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες αυτές. Και τέλος οι προφορίες ε, που, και οι συμβουλές που γίνονται, προ του προς τους μέσω του ιστοσελίδα HOA. Ποιες είναι οι προοπτικές λοιπόν για το μέλλον. Στο άμεσο μέλλον μπορούμε να προβλέψουμε μια, μια αύξηση των ε, επιθέσεων μετά το πέρα των μουσώνων και το 2010 οι ε, συνεισφορές των κρατών μελών θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουν δίχως καμία δυσκολία η επιχείρηση αλλά η εκρίζωση της πειρατείας θα παραμείνει αδύνατη εάν δεν ε, ασχοληθούμε με την ουσία του προβλήματος και τις βασικές αιτίες. Γι' αυτό λοιπόν αφήσαμε να ε, ξέρουμε μια ανέστακη για την Σομαλία. Στον στρατιωτικό τομέα έχουν οριστεί τρεις ε, τομείς, ε, την ενίσχυση της Ινισόμ, την που υποστηρίζει με 5.000 άνδρες ε, την προσωρινή κυβέρνηση να υπάρξει στρατιωτική συνεργασία βοηθώντας ε, τις ε, παράκτιες χώρες του Ινδικού ωκεανού να λάβουν έλεγχο της περιοχής και να υποστηρίξουμε, να βοηθήσουμε τις, σωμα, τις δυνάμεις της Σομαλίας. Αυτή τη στιγμή προπαρασκευάζονται οι προτάσεις οι οποίες ε, θα υποβληθούν από το Συμβούλιο. Όπως ξέρετε, συμμετέχουμε σε διάφορα συμβούλια για την βοήθεια στην Αφρική ε, σχετικά με την διατήρηση της ειρήνης ε, στο Κονγκό για την μεταρρύθμιση των στρατιωτικών δυνάμεων αλλά και των αστυνομικών δυνάμεων και στη Βουλή Μπισάου να, θα φροντίζουμε να το πράξουμε εάν μας το επιτρέψει το περιβάλλον. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στις ικανότητες της θεωρητικής μας, είναι η προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας ε, και οι στόχοι είναι τρεις. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ε, δυνατότητας χρήσης των, ε, των μάχημων ομάδων, να αυξήσουμε την, ναυτική μας ε, συμμε... ναυτική συμμετοχή με μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των κρατών και να φροντίσουμε για μια καλύτερη διαχείριση των κρίσεων τώρα επί των θεμάτων αυτών και την κατάργηση των ελλείψεων και των ανεπαρκειών που έχουμε η Στρατιωτική Επιτροπή ε, συνεργάζεται συχνά με την ε, Επιτροπή Άμυνας στην περίοδο αυτή τη οικονομική κρίση θα πρέπει να τονίσω ότι οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για τι αποστολέ στο εξωτερικό σπανίζουν όλοι οι προπολογισμοί άμυνας των Ευρωπαϊκών κρατών βρίσκονται σε πτώση, φθήνουν και οι κρίσει που πλήττουν τι πιο φτωχέ χώρες δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν νέε εντάσεις και νέα βία. Πιστεύω προσωπικά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το αγνοήσει ε, διαφορετικά όλα αυτά θα αποβούν εις βάρος της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε ε, στρατηγέ για αυτή την πολύ πλήρη αλλά και σύντομη ε, παρουσίαση που μας δίνει δυνατότητα να συζητήσουμε. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις που προβλέπονται. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Βανόρντεν και θα παρακαλέσω βέβαια να είστε αρκετά σύντομος στις παρεμβολές σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα το να σας βλέπω σε αυτή την Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι πολλοί από εμά έχουν ορισμένες δυσκολίες να ε, κατανοήσουν την αρχή της ΕΠΑ, η οποία είναι ουσιαστικά μια ένα πολιτικό επιχείρημα. Ε, ε, πολλά από αυτά τα θέματα έχουν σχέση με το ΝΑΤΟ και ζητήσαμε να υπάρχει ένα ε, ευρωπαϊκό μια ευρωπαϊκή προσπάθεια που να επηρεάσει την κατάσταση. Βλέπω ότι εντασσόμαθε τώρα και στην στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ. Πώς προβλέπετε τη μελλοντική συνεργασία και ιδίω πώς θα συνεργαστούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί σε μια περίοδο οικονομικής στενότητος όπου όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους και πάσχει και η άμυνα από αυτό παρόλες τις σοβαρές δυσκολίες που έχουμε όταν ε, πρόκειται για σειρά ξανά τον κόσμο και το παρακολουθούμε ε, υπάρχουν δύο οργανώσεις οι οποίες και αυτές ιδίω αποτελούνται από συστατικά ευρωπαϊκά και μάλλον ε, συναγωνίζονται στον ίδιο χώρο. Αντιλαμβάνομαι τις διαφορές τις οποίες αναφέρατε, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά την κατανομή των δυνάμεων μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό σκέλος. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα με το οποίο κατέληξε ο κύριος Βανόρντεν είναι κάτι που και εγώ θέλω να θέσω ιδίω ε, και αν δεν συμφωνώ με όλες τις απόψεις τους, παραδείγματος χάρη για το Αταλάντα και ε, το παραλληλισμό του, ε, με το ΝΑΤΟ και το πρόγραμμα Ocean Shield που υπάρχει στις ακτές της Σομαλίας. Γιατί δηλαδή η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ επιχειρούν στον ίδιο χώρο δύο διαφορετικές ε, ε, δραστηριότητες. Πώς οργανώνεται δηλαδή αυτό. Έχω όμως επίσης ε, και άλλα ερωτήματα, διότι κύριε στρατηγέ τελειώνει τώρα η δραστηριότητα σας και ε, ίσως ε, είναι διαφορετικές τώρα οι απόψεις σας από το What Aspiration for European Defense το οποίο έχω διαβάσει διότι αναφέρεται την ανάγκη αναδιοργανώσεως της Γενικής Γραμματείας της Βρυξέλλες για τη διαχείριση των κρίσεων. Δηλαδή σε ποιες εμπειρίες βασίζεστε στα πλαίσια της ΕΠΑ για να καταλήξετε σε αυτές τις συστάσεις. Έχω και άλλη μία ερώτηση όσον αφορά τον ε, στόχο ο της Γαλλικής Προεδρίας ε, στην ε, ε, προηγούμενη χρονιά είχαν παρουσιαστεί οι προβλεπόμενες δυνάμεις και υπήρχε η διακήρυξη για την ενίσχυση των δυνάμεων του τέλους του 2008 όπου αναφέρατε 60.000 άτομα που θα μπορούν να κινητοποιηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, και καλυμμένοι ή ρητοί αυτοί οι στόχοι θα μπορέσουν να επιτευχθούν σύντομα και είναι σωστό να έχουμε δύο προγράμματα τα οποία ε, ε, έχουν παράλληλα, δηλαδή τα e-battle groups και οι κινητές δυνάμεις. Αυτές είναι οι πρώτες μου ερωτήσεις για, σαν εισαγωγή και θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέμκε. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση διότι είσαστε ε, πολύ έμπειρος και ίσως είναι αντιφατικά αυτά που θα σας πω, αλλά αναφερθήκατε σε αποστολές και στρατιωτικές και παρατηρητικές. Και θα ήθελα να σας πω ότι εφόσον προέρχομαι από μία χώρα η οποία δεν έχει συμμετάσχει ούτε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, ούτε σε αποστολές παρακολούθησης σε στρατιωτική περιοχή, γίνεται. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ε, θα ήθελα να ξέρω τι ε, γίνεται με τις διάφορες επιτροπές διότι εάν από τον Ιανουάριο υιοθετηθεί η συνθήκη της ε, Λισαβόνας έχετε σκεφτεί ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για ε, το, τη δικιά σας δύναμη από την υιοθέτηση της συνθήκης αυτής όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Ευχαριστώ. Προτείνω να απαντηθούν αυτές οι πρώτες ερωτήσεις και μετά θα υπάρξουν νέες δύο ομάδες των τριών ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, είναι χαρά μου που έρχομαι εδώ γιατί τουλάχιστον δεν είναι επουσιώδεις οι ερωτήσεις οι οποίες τίθενται όπως καμιά φορά συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δηλαδή αν αυτά τα οποία κάνουμε εξυπηρετούν κάποιο στόχο. Εάν δηλαδή στην πραγματικότητα ό,τι γίνεται στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας δεν θα γινόταν καλύτερα από το ΝΑΤΟ, το οποίο εξασκεί αυτά τα καθήκοντα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πιστεύω για να μην σας κρύψω τίποτα εφόσον ε, είμαι απερχόμενος ότι με υποψιαζόταν το επιτελείο μου στο Παρίσι ότι προτού αναλάβω αυτά τα καθήκοντα ήμουν ευρωσκοπητικιστής και γι' αυτό δεν ήμουν δογματικός. Ήρθα εδώ με το συνέστημα ότι μπορούσαμε κάτι να κάνουμε το συγκεκριμένο και όχι μόνο έχω έχω πιστεί, αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάνουμε έχει κάποια σκοπιμότητα και χρησιμότητα. Και θα είμαι συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συναγωνίζονται και ε, ε, αυτός ο ανταγωνισμός είναι εις βάρος και των δύο. Ατυχώς καμιά φορά ναι, αλλά θα σας έλεγα ότι αυτό οφείλεται περισσότερο στις νοοτροπίες και στα πολιτικά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο οργανώσεων που όλοι γνωρίζετε και δεν θα επεκταθώ και λιγότερο σε μία πραγματική στρατιωτική ε, ε, ανταγωνιστικότητα διότι ε, όπως ξέρετε οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο οργανώσεων είναι συνεχείς. Ο Ιταλός ομόλογός μου στο ΝΑΤΟ είναι ένας παλιός μου φίλος και συναντιόμαστε πολύ συχνά και τηλεφωνιόμαστε μόλις προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αντιθέτως, ε, τι κατάρτιση εργασιών μπορεί να γίνει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ. Είναι αρκετά απλό. Ε, υπάρχει μία πρώτη περίπτωση την οποία διαπιστώνουν στο Κωσυφοπέδιο και στο Αφγανιστάν όπου το ΝΑΤΟ ε, ε, έχει τις στρατιωτικές δυνάμεις και η ΕΠΑ έχει τις, τους οικονομικούς πόρους και επιβαρύνεται και με την πολιτική αποδομή. Επίσης οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο οργανών αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες όπως το υπενθύμισε ο κύριος Ράσμουσεν. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι καλή αυτή η συμπληρωματικότητα και ένα δεύτερο στοιχείο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε καλύτερη θέση από ότι το ΝΑΤΟ για να προβεί στην πρόληψη ε, μίας κρίσεως που δεν δεν είναι ε, μεγάλη σύραξη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες ε, συγκρούσεις ε, και γι' αυτό δεν έχει συμφωνηθεί για κάτι τέτοιο στην συνάντηση του Πέτερσμπεργκ. Μπορούμε λοιπόν, δεν μπορούμε λοιπόν μόνοι μας να αναλάβουμε τη διαχείριση της κρίσης, το είπα προηγουμένως και για το Τσάντ. Δηλαδή οι ε, αντιμαχόμενες δυνάμεις είτε πρόκειτο για το Τσάντ είτε για το Σουδάν δεν θα δεχόντουσαν να υπάρξει μία δύναμη του ΝΑΤΟ η οποία θα επενέβαινε ούτε του ΟΗΕ. Άρα αυτό το οποίο κάναμε για τις 420.000 προσφύγων στο Τσάντ που ήταν κάτι που δεν μπορούσε να κάνει κανείς άλλος πλην ημών. Με συγχωρείτε, ε, ε, κλείνω το ένα μικρόφωνο. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εκεί από πιο παλιά και γι' αυτό το λόγο έχει τη δυνατότητα να συντονίσει και τις πολιτικές και τις στρατιωτικές δυνάμεις και γι' αυτό είναι πιο αποτελεσματική και αυτό ισχύει για το πρόγραμμα Αταλάντα διότι όταν οι Ευρωπαίοι χρειάστηκε να ε, να δώσουν τις ε, δυνατότητές τους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση τα, τα στρατιωτικές δυνάμεις αποφάσισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερα καταρτισμένη για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα και νομικά και οικονομικά από ότι το ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός με το ΝΑΤΟ, απλούστατα έχω προσπαθήσει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια γιατί από πλευρά στρατιωτικής δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε ακριβώς όλους τους κανόνες και όλες τις ιδέες και να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι πρόκειται να κάνουμε ε, και οι δύο πλευρές. Γιατί λοιπόν ε, σήμερα ε, δύο επιχειρήσεις συγκεκριμένα Σομαλία κατά της πειρατείας, εγώ ε, λυπούμαι γι' αυτό πρέπει να σας πω προσωπικά. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πρώτη επιχείρηση ήταν μια ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία έγινε εκεί. Και είναι προφανές ότι η επιφάνεια 3.000 ε, χιλιόμετρα της Σομαλίας είναι τόσο μεγάλη που όσο περισσότερα πλοία είναι εκεί τόσο το καλύτερο. Όταν αρχίσαμε λοιπόν να ζητούμε από το ΝΑΤΟ να εμπλακεί εγώ συμφώνησα ε, να συμμετέχει και το ΝΑΤΟ εφόσον ούτε η Τουρκία ούτε ε, οι, οι, Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό στόλο και μπορούσαν να αναπτύξουν εκεί στόλους. Η SNMG η οποία βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του ΝΑΤΟ έχει μόνο 3-4 πλοία τα οποία όμως είναι μια σημαντική προστιθέμενη αξία αποτρεπτική ε, όσον αφορά την ανθρωπιστική ψυχή και ε, την ε, στήριξη. Όσον αφορά τις απόψεις του Συμβουλίου, εγώ δεν μπορώ εδώ ε, να αναφερθώ διότι δεν εντάσσεται με, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ εδώ και τρία χρόνια από όταν εγώ ενεπλάκην. Δηλαδή, αν ε, υπήρχε όλο και μεγαλύτερη ε, ε, συνένωση των πολιτικών και των στρατιωτικών σκελών. Δηλαδή όσον αφορά τις πληροφορίες πολιτικές και στρατιωτικές. Εμείς συνεργαζόμαστε πλήρως με το intelligence του επιτελείου. Επίσης όσον αφορά την παρακολούθηση υπάρχει πλήρη συνεργασία των πολιτικών με και των στρατιωτικών δυνάσεων. Το CPCC επίσης έγινε με μόνιμη στήριξη του επιτελείου όλου του προγραμματισμού των πολιτικών ε, επιχειρήσεων. Παραδείγματο χάνει για τη Γεωργία είχαμε αποσπάσει πέραν του ενός μήνα ε, εις ε, τη δύναμη αυτή 17 αξιωματικούς του επιτελείου οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά εις τα θέματα αυτά. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη αρκετά διότι όπως ξέρετε ένας από τους στόχους της Γαλλικής Προεδρίας ήταν να υπάρχει μία πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία με πλήρη ε, ένταξη, πράγμα το οποίο δεν έχει ακόμη ε, υλοποιηθεί και για μένα θα αποτελέσει ένα βασικό ε, θέμα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εφόσον δεν ε, έχουμε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, δεν έχουμε ούτε τη μεγάλη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ, ούτε την εμπειρία της στρατιωτικής ε, ε, αρχηγίας του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών δυνάμεων. Πού βρισκόμαστε τώρα σχετικά με τη δύναμη των 60.000 ατόμων. Όντως η Γαλλική Προεδρία είχε προτείνει αυτό το οποίο ορισμένοι είχα θεωρήσει σαν ένα νέο ε, επίπεδο φιλοδοξιών. Ο στόχος όμως αυτός υπάρχει από την αρχή. Δηλαδή, αυτό είχαμε διαπραγματευτεί από ε, από το έτος 2000. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι νέο. Αυτό που είναι νέο είναι η επιμονή του εγγράφου αυτού το οποίο να απεδέχθη το Συμβούλιο. Δεν είναι δηλαδή πλέον μόνο ένα γαλλικό έγγραφο για την υποχρέωση εντός 10 ετών γιατί ήμασταν επιφυλακτικοί να υπάρξει υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να κινητοποιήσει αυτές τις 60.000 ε, στρατιώτες ε, για διάφορες ε, επιχειρήσεις που διεξάγονται συγχρόνως. Όλα αυτά λοιπόν είναι φιλοδοξίες και υποθέσεις εργασίας αλλά βεβαίως αυτό δεν εγγυάται ε, καμία στιγμή ότι θα μπορέσουμε ε, να έχουμε στη διάθεσή μας τους πόρους και ότι θα μας τους διαθέσουν οι κυβερνήσεις. Για το Τσάντ και την Κεντρική Αφρική χρειαστήκαμε έξι μήνες για να μπορέσουν να συγκεντρώσουμε 3.700 άτομα τα οποία χρειαζόμασταν. Αν βλέπαμε τον κατάλογο των δυνάμεων που αναφέρεται σε 60.000 άτομα θα λέγαμε βεβαίως έχουμε τις αναγκαίες Οπότε αυτό το επίπεδο των φιλοδοξιών είναι απλώς θεωρητικό στόχος που μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε, να βελτιώσουμε τις δυνατότητες μας, αλλά όχι μια μεγαλύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχει σήμερα ένα κράτος μέλος το οποίο δεν συμμετείχε σε τίποτα ε, πιστεύω ναι, αλλά δεν είμαι βέβαιος και δεν έχω ψάξει. Αλλά τα τελευταία τρία χρόνια οι ιδέες έχουν αλλάξει. Όταν εγώ ξεκίνησα σε αυτή την στρατιωτική εμπλοκή, είχα ως επτοπλίστων απέναντί μου τους αρχηγούς των επιτελείων που ήταν και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φέρναν και τα δύο καπέλα και αυτό που του ενδιαφέρε ήταν το καπέλο του στο ΝΑΤΟ και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι τώρα υπάρχει μία συλλογική ε, προοδευτική ε, εξέλιξη και για το Τσάτ και για την Αταλάντα είδαμε ότι έχουν αλλάξει ιδέες. Δηλαδή τώρα ένας στρατιωτικός εγκαταλείπει τη θέση του μετά από τρία χρόνια και αποχαιρετά τους ομολόγους τους. Δεν ακούει πια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονιστεί περισσότερο με τον ΝΑΤΟ διότι διαπιστώνουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε επίσης να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε κάτι. Άλλαξαν λοιπόν οι ιδέες και αν ακόμη σήμερα υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν σε καμία επιχείρηση, όλο και περισσότερες χώρες συμμετέχουν σε κάθε νέα επιχείρηση και σε δύο-τρία χρόνια πιστεύω ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης θα, συμμε... θα έχουν συμμετάσχει σε μία επιχείρηση. Όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορώ να σας πω απολύτως τίποτα, διότι έχουμε ε, λάβει σαφείς οδηγίες από τον Ξαβιέ Σολάνα και θέλω να τη σεβαστώ. Δηλαδή ε, όσο δεν έχει κυρωθεί η συνθήκη δεν πρόκειται να επεκταθούμε καθόλου επ' αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ε, το να είσαστε τόσο ο εκτενής στα περισσότερα θέματα, ο κύριος Γιάννης Μπάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και να καλωσορίσω τον ε, στρατηγό Ζαντ και τον ευχαριστώ επίσης για την εξαιρετική ομιλία του και τις απαντήσεις που έδωσε στους ε, συναδέλφους τις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Θα ήθελα να πω τώρα για την ΕΠΑ ότι μέσα σε πολύ μικρό διάστημα κατόρθωσε να πετύχει μία σειρά στόχων και να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο που αν σκεφτούμε πως πρόκειται μόνο για 5-6 χρόνια αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπήρχαν και κάποια κράτη, μην ξεχνάμε, που ανθίσταντο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αναφερθήκατε στην προσθεμένη αξία σχετικά με τα όσα ειδοποίησε η ΕΠΑ. Φυσικά είχε κάποιους περιορισμούς θεσμικού χαρακτήρα και μετά από τις οδηγίες του συμπατριώτη μου κ. Σολάνα η ΕΠΑ θα αποτελέσει την ραχοκοκαλιά για μια μελλοντική πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, ουσιαστικότερη στην Ευρώπη. Ε, ο επικεφαλής ε, της, ε, του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές στην Ιαπωνία είχε πριν από τις εκλογές προσπαθήσει να αξιολογήσει και να περιγράψει το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και εξέφρασε το θαυμασμό του. Επαναλαμβάνω λοιπόν πως ε, ε, η σπονδυλική στήλη της ΕΠΑ είναι η ε, ευρωπαϊκή πολιτική, η εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική. Και ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με την Αταλάντη. Αναφερθήκατε στην ε, συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στην επιχείρηση Αταλάντη. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην, η ερώτηση να είναι δική της, δική της αρμοδιότητας, αλλά το γνωρίζετε. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία μόνο και μόνο κυνηγώντα ε, τους πειρατές. Χρειάζεται και κάτι άλλο. απαιτείται να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται τα τεράστια ποσά των λίτρων. Μόνο έτσι λοιπόν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την πειρατεία στην Σομαλία και στον Ινδικό ωκεανό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκαλτιέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον στρατηγό για τις εργασίες του τα τελευταία χρόνια και για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ε, και εξήγησε ότι αυτές οι ιδιαιτερότητες ε, βρίσκονται στην βάση της επιτυχία της, ε, το οποίο προκύπτει και από τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία πολλές φορές θεωρείται ως ένας ε, πολύ αξιόπιστος εταίρος και πολύ επισημητός θα έλεγα. Και φυσικά όπως βλέπουμε υπάρχει και μια ανάμειξη σε, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο στρατιωτικό. Από το 2003 λοιπόν θα έλεγα είχε ξεκινήσει ουσιαστικά η ΕΠΑΕ η οποία τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε, αναπτύχθηκε περαιτέρω και θα πρέπει να συνδυαστεί περισσότερο κανένα με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Τώρα είχαμε μια σειρά επιτυχιών της ΕΠΑ αλλά αυτά, αυτές οι επιτυχίες έχουν καταδείξει κάποια όρια. Υπάρχει λεγόμενη κρίση οφειλόμενη στην ανάπτυξη. Τώρα υπάρχει το ζήτημα των στρατιωτικών ε, ικανοτήτων. Ακούσαμε τους ε, στόχους της Γαλλικής Προεδρίας που ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξοι. είναι κάτι που τόνισε πρόσφατα και το Συμβούλιο. Ακούσαμε τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας και θέλω να ακούσω από τον στρατηγό ποιο είναι το βασικό πρόβλημα των στρατιωτικών ε, ικανοτήτων που αφορούν πρωτίστως ε, τα ελικόπτερα και την αξιοπιστία και λειτουργία ε, έχω χαρακτήρα αυτού του προγράμματος που είναι μέσω μακροπρόθεσμο και τις δυνατότητες που έχει το πρόγραμμα αυτό να εκμεταλλευτεί όλες τις ευρωπαϊκές δυνατότητες που προσφέρει η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αγορά ελικοπτέρων, σε ό,τι αφορά την α400 μη. Θα ήθελα να αναφερθώ στους ε, μάχημες ε, στρατιωτικές ομάδες ε, τακτικής τις τακτικές ομάδες και την άμεση απάντηση, άμεση ανταπόκριση. Και τώρα θα ήθελα να θίξω κάποια αισθήματα που αφορούν την συνθήκη της Λισαβόνας, το ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα στην ε, στρατιωτική διάσταση και την πολιτική διάσταση και θέμα της αξιολόγησης με καλύτερο τρόπο αυτό το σώμα, του σώματος που ε, απεικονίζει καλύτερα την, ε, το ζήτημα αυτό, δηλαδή της ε, ευρωπαϊκής χωροφυλακής και το πώς μπορεί να επιτευχθεί ένας καλύτερος συντονισμός τόσο στην βάση όσο και στην κορυφή. Να μην λοιπόν είναι υπεύθυνο μόνο ο επιτόπου ύπαρος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, κύριε Βανμπάλεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ρωτήσω το στρατηγό το εξής. Στη συμμετοχή της ΕΠΑ από το Πίτερσπουργκ μέχρι το Σεν Μαλό και παραπέρα, βλέπουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε ολόκληρο το στρατιωτικό φάσμα. Οι επιχειρήσεις όμως συνήθως ε, γίνονται ε, ε, στο ήπιο φάσμα του στρατιωτικού σκέλους, ειρηνευτικές κλπ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, ασκώντας μεγαλύτερη διεθνή επιρροή, πρέπει να μπορεί να είναι έτοιμη να κάνει και ε, μεγαλύτερης κλίμακας ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Είμαστε εξοπλισμένοι για κάτι τέτοιο. Ξέρω βέβαια ότι ε, ε, ε, είστε βέβαια δημόσιος υπάλληλο, αλλά πιστεύετε ότι υπάρχει αυξημένη πολιτική βούληση ούτω ώστε να λάβουν χώρα και τέτοιου είδους μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο κ. Κουμούτσακος, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον στρατηγό για την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Στρατηγέ, όπως είπατε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, η SDP, παρά το γεγονός ότι είναι νεαρή σε ηλικία, έχει ήδη να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό απολογισμό. Και στη βάση αυτή νομίζω ότι όλοι έχουμε την αισιοδοξία και την προσμονή και έχουμε λόγο να αισιοδοξούμε ότι και με την θέση σε ισχύ της Λισαβόνας, της συνθήκης Λισαβόνας, οι προοπτικές της ESDP θα είναι ακόμα καλύτερες στο μέλλον. Και επειδή ακούστηκε ποιος θα είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία ή ποιο είναι το κριτήριο κατανομής ρόλων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η SDP και ΝΑΤΟ, εδώ αρκεί καλής να αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις ασφάλειας ή οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων συνήθως γίνονται σε περιοχές που δυστυχώς ή ευτυχώς οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες δεν είναι τόσο θετικές για την παρουσία της νατοικής σημαίας σε αυτές τις περιοχές. Αντιθέτως υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή και σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και σε επίπεδο πολιτικού περιβάλλοντος για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά κριτήρια που κανείς θα μπορούσε να αναφέρει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και ποιες είναι προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας απαιτεί από την SDP μεγάλες προσαρμογές, προσαρμοστικότητα. Και μία από τις σύγχρονες απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι τα μεγάλα κύματα λαθρομετανάστευσης τα οποία αντιμετωπίζουμε ως φαινόμενο και περιφερειακών κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό βεβαίως υπάρχουν ήδη δομές όπως η Frontex κτλ. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να έχω ένα σχόλιο, μια σκέψη στο ενδεχόμενο στο πλαίσιο της Frontex ή αυτής της στρατηγικής στο μέλλον να διαμορφωθεί και να συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή μια δύναμη ευρωπαϊκής Ακτοφυλακή. Γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται μαξιμαλιστικό αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι πεπισμένο ότι το μέλλον της ESDP βασίζεται σε πρωτοποριακέ και μαξιμαλιστικέ ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ, κύριε Στρατηγέ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για το πρώτο σημείο, σας φυσικά για όλα τα σχόλια που κάνατε και με τα οποία συμφωνώ απολύτως, όταν ε, θίξατε το θέμα της ε, συμπληρωματικότητας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Φυσικά δεν φέρουμε τις ίδιες ευθύνες. Ε, το ΝΑΤΟ ασχολείται με την συλλογική άμυνα. Κάτι το οποίο σημαίνει και περισσότερα μέσα, περισσότερα στρατηγία κλπ. Αλλά όταν βλέπουμε τα πράγματα από την πλευρά της διαχείρισης των κρίσεων, χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι σε ό,τι φορά το κόστος αποτελεσματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει πολύ καλά. Η στρατηγική δομή του ΝΑΤΟ, γι' αυτό και θα μιλάμε η επικάλυψη, με κάνει μερικές φορές να χαμογελάω, η στρατηγική δομή λοιπόν του ΝΑΤΟ εκπροσωπεί σήμερα 15.000 άτομα και η ευρωπαϊκή δομή αποτελείται από 200 άτομα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα αυτό κατά νου. Τώρα, η Αταλάντη, τι να κάνουμε, ειδικά σε ό,τι φορά το οικονομικό κύκλωμα, κανείς δεν αγνοεί πως αν η πειρατεία διατηρείται και εξελίσσεται, αναπτύσσεται, οφείλεται στο ότι οι αλείς ε, έχουν κάθε συμφέρον. Γιατί πρόκειται για αλληλείς στην ουσία. Εντάξει, υπάρχει ένα κύκλωμα μέσα στο οποίο κυκλοφορεί το χρήμα, τα λίτρα, κάτι το οποίο αρχίζουμε να μαθαίνουμε. Οι Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν μια ομάδα επαφής ε, στο πλαίσιο της οποίας ε, κράτη με, ευρωπαϊκή, συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ δραστήριες και ενεργές και αυτή η ομάδα επαφής ανέθεσε σε μια ομάδα εργασία να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Η ομάδα αυτή εργασία φυσικά αντιμετωπίζει πάρα πολλά εμπόδια. Κάθε φορά όταν ε, υπάρχουν διεθνή οικονομικά κυκλώματα, πολλά κράτη δεν ε, είναι υπέρ της ε, ανάμειξης στα εσωτερικά τους οικονομικά κυκλώματα κλπ τραπεζικό απόρριτο και άλλα. Τώρα, ε, περισσότερη ανάπτυξη της ε, ΑΕΠ, της ε, ΕΠΑ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε να λάβουμε μια νέα επιχείρηση, αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. τώρα, το, τα ζήτημα των ελικοπτέρων, το πρόγραμμα προχωράει. Ξέρετε ότι είναι ένα κοινό πρόγραμμα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι που σπανίζει, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όντως προχωράει. Αλλά προς το παρόν είναι περιορισμένης εμβέλειας που πρέπει να αντιμετωπίσει προς το παρόν τις άμεσες ανάγκες και την ε, στοχεύει στην ανακύκλωση ορισμένων ελικοπτέρων και πληρωμάτων ρωσικής προέλευσης ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο σύνολο των θεάτρων, των επιχειρησιακών θεάτρων. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία ξεκινάνε και φαίνεται πως έχουν κάποιο μέλλον. Τόσο φορά το Airbus 400M, οι Υπουργοί Άμυνα ε, αποφάσισαν να δώσουν μια νέα ευκαιρία στο πρόγραμμα αυτό και πρόκειται να συνενεθούν σε μερικούς μήνες για να δουν πώς προχωράει ο φάκελος αυτός ε, αλλά και την ε, δυνατότητα υποβολής νέων προτάσεων από την ε, αεροναυπηγική εταιρεία. Αυτά, που ξέρετε, είναι θέματα που δεν ε, απασχολούν άμεσα την δική μας Επιτροπή τώρα σε ό,τι φορά το Battle Groups, τις μάχες ομάδες και τις ομάδες ταχείας ανάπτυξης. Αυτή είναι μια από τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτά τα Battle Group. Για ποιο λόγο, αυτό είναι το ερώτημα που έχουν θέσει και οι Σουηδοί, είναι ένα ζήτημα επί του οποίου εργαζόμεθα. Αυτά τα battle group δεν ε, χρησιμοποιούνται επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα φανταστικό, εικονικής ε, πραγματικότητας κλπ. Έχουν κάποιες ε, ελλείψεις, έχουν ελλείψεις στερεωτικών ικανοτήτων ή δυνατοτήτων γεγονό είναι ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο, διότι και πιστεύω πω πολλά πρέπει να βελτιωθούν. Είμαι αισιόδοξο, διότι θεωρώ ότι πρόκειται για πολιτική βούλη στην ουσία. Ότι δηλαδή για να χρησιμοποιήσουμε μια δύναμη ταχεία ανάπτυξη είτε του ΝΑΤΟ είτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται το σύνολο των κρατών να συμφωνούν. Και για να συμφωνήσουν 27 χώρε για να ε, χρησιμοποιηθεί ε, λιγότερο από 15 μέρες μία ε, μάχη, μία ομάδα, τότε το ζήτημα θα πρέπει να είναι ζωτική σημασία για όλους. Πιστεύετε ότι κάτι θα συμβεί. Δεν το πιστεύω, διότι στη Γεωργία αποδείχθηκε το αντίθετο. Εντάξει, πρόκειται για μια αποστολή πολιτικού χαρακτήρα, θα λέγαμε, αλλά χρησιμοποίησαμε ως επιτοπλίστων την χωροφυλακή. Η ανάπτυξη λοιπόν έγινε διότι όλοι συμφώνησαν πως ε, η περίπτωση ήταν επίγουσα, ζωτική σημασία κλπ. Και θα ξανασυμβεί όταν κρίνουν κάτι το παρόμοιο στο μέλλον. Τώρα, το ζήτημα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Χωροφυλακής, εργαζόμαστε πάνω σε αυτό για την Βοσνία, διότι σήμερα το η χωροφυλακή η οποία βρίσκεται εκεί έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Χωροφυλακή αλλά όπως ξέρετε δεν ε, έχουμε αποστείλει μόνο εκεί τέτοια ομάδα αλλά και στο Αφγανιστάν. Τώρα για τις ε, πολιτικές επιχειρήσεις ε, ένας η δυνατή, θα αποτελέσει την καλύτερη δυνατή απάντηση σε κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα. Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σήμερα βρίσκονται σε χαμηλό βαθμό, χαμηλό επίπεδο, μπορούμε να στοχεύσουμε πιο ψηλά. Μπορούμε να σκεφτούμε επιχειρήσεις ε, είδους ε, ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Η απάντηση σήμερα είναι όχι. Για να είμαι πραγματικά ειλικρινής, το πρόβλημα που υπάρχει για μας από στρατιωτική σκοπιά είναι ότι μια επιχείρηση όπως το Αφγανιστάν ή το Ιράκ είναι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ε, γίνουν χωρίς την συμμετοχή των ΗΠΑ και είναι μάλλον αδύνατο να συμμετάσχουν οι Αμερικανοί και να ενταχθούν σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Σήμερα όπως έχουν τα πράγματα αυτό αποκλείεται. Ίσως κάποτε να συμβεί στο μέλλον. Διότι τέτοιες επιχειρήσεις ε, απαιτούν την συμμετοχή των Αμερικανών και στην περίπτωση αυτή μόνο το ΝΑΤΟ μπορεί να αναλάβει τέτοιες επιχειρήσεις ε, επιχειρήσεις δηλαδή μεγάλου ελληνικού ε, οι ικανότητες πληροφοριών και διοίκησης δεν επαρκούν για τέτοιες επιχειρήσεις μεγάλου ελληνικούς. Είχαμε μια επιτυχή ε, επιχείρηση στο Τσάντ και στην Κυριακή Αφρική πάνω σε ε, θέμα εχθρικό περιβάλλον κλπ. Ε, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Αυτό δείχνει ότι έχουμε τις δυνατότητες αλλά για ε, περιπτώσεις και επιχειρήσεις μικρότερες ευέλειες. Εάν λοιπόν βρεθούμε σε μια περιοχή όπως το Αφγανιστάν, τώρα θα χρειαστούμε περισσότερες ε, ικανότητες ε, και δυνατότητες ε, τόσο επίπεδο πληροφοριών όσο και σε επίπεδο διοίκησης τώρα. Κατά πόσο χρειάζεται τώρα ένα ε, στρατηγείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει συζητηθεί επανειλημμένα και τα κράτη-μέλη είναι διχασμένα. όταν συζητώ με τους ε, αρχηγούς ε, των επιτελείων. Υπάρχει μια κάποια πλειοψηφία που θεωρεί ότι ναι πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό στρατηγείο, υπάρχει μια μειοψηφία που θεωρεί πως όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο και δύσκολο. Όσοι επιθυμούν το στρατηγείο μιλάνε για αποτελεσματικότητα, στρατηγική, πολιτικοστρατηγική κλπ. Και οι υπόλοιποι λένε πως ο κίνδυνος θα είναι εάν υπάρξει ένα ευρωπαϊκό στρατηγείο θα δημιουργήσουμε έναν ανταγωνισμό με το ΝΑΤΟ και αυτό θα επηρεάσει τις Διατραντικέ μας ε, σχέσεις. Ε, λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει ε, γενική συμφωνία και πλήρη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων για να, να συσταθεί ένα τέτοιο στρατηγείο, το ζήτημα δεν τίθεται καν. Τώρα, οι επιχειρήσεις στις περιοχές της μειονεκτούσες, παράνομη μετανάστευση και κλπ. Μετανάστευση. Τώρα αυτό ξεπερνάει το θεωρητικό πλαίσιο διότι είναι κάτι ε, το οποίο αφορά όπως αναφέρατε την Κομισιόν και ιδιαίτερα το Frontex. Φυσικά εμείς δεν ε, αδιαφορούμε διότι στη συντριπτική πλειοψηφία είναι οι εθνικές ε, ναυτικές δυνάμεις που συμμετέχουν. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν της λάθρομετανάστευσης ε, συνδυάζεται με ένα πρόβλημα εμπορίας ναρκωτικών, ε, υπάρχει ζήτημα τρομοκρατίας ε, κλπ. Ένας από τους βασικούς στόχους της Οδικής Προεδρίας είναι να προωθήσει την εποπτεία των θαλασσίων συνόρων, διότι εδώ χρειάζονται φυσικά εκτός από τα ναυτικές δυνάμεις και αεροπορικές δυνάμεις κλπ. Και θα πρέπει μονίμως και συνεχώς να εποπτεύουμε τις, τα θαλάσσια σύνορά μας γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά πρέπει να γίνουν, πολλά να γίνουν και σε συνδυασμό και συντονισμό με τον ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ε, ζήτησε τις υπηρεσίες πέντε ναυάρχων οι οποίοι θα αναφέρουν ε, προσεχές έτος ε, σε εκθέσεις τους, ε, το, τις που υπάρχουν για το ναυτικό μας έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα ε, σήμερα μεταξύ της ε, πολιτικής και στρατιωτικής ΕΠΑ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, και πρέπει να δοθεί έμφαση και στα δύο σκέλη. Είπατε ότι δουλεύετε πάνω σε αυτό το θέμα, μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις, μπορείτε να το εξηγήσετε πώς θα υπάρχει αυτή η συνεργασία. Επίσης είχα τη δυνατότητα να πάω στη Γεωργία και να δω την αποστολή επιτόπου. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετέσχουν σε αυτή την αποστολή ε, πολύ γρήγορα αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις σε δύο εβδομάδες στη Γεωργία. Ήταν καταπληκτικό το επίτευγμα και σε σχέση με τη Σομαλία. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπαίνει ένα θέμα εφοδιασμού όταν αναπτύσσονται γρήγορα δυνάμεις ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε για να υποστηρίζεται σωστά το προσωπικό. Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν λοιπόν ούτως ώστε ο ανεφοδιασμός να γίνεται και, και η επιμελητία να γίνεται όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ο στρατηγός Μπεντεζά έχει πιο περιορισμένο χρόνο από ό,τι πίστευα, οπότε παρακαλώ οι πέντε επόμενοι παρεμβαίνοντες να περιοριστούν σε μία ερώτηση για να έχουμε μία τελευταία ανταλλαγή. Ο κύριος Έρενχάουζερ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ε, ε, αλλά είχα τέσσερις ερωτήσεις. να κάνω, θα, ρωτήσω, θα κάνω τη μία μόνο. Είπατε ότι η υπηρεσία πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε πολύ τον τελευταίο καιρό. Κυρίω ε, ενσωμάτωσε και τον πολιτικό τομέα, οπότε θα σημαίνει αυτό ίσως ότι ε, έχει διαλυθεί η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ε, ή πώς εννοείται την ενσωμάτωση με τον πολιτικό τομέα της υπηρεσίας πληροφοριών. Ευχαριστώ. Η κυρία Λιουζινγκ. Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δόθηκε να κάνουμε ερωτήσεις σε ένα υψηλό βαθμό στρατιωτικό στέλεχος. Στην αρχική σας δήλωση είπατε ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση επέδρασε δυσμενέστατα ε, στις... Ε, ε, χώρες και μπορεί να ε, υπάρχουν προβλήματα και για την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω μήπως υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια που έχετε κατά και αν υπάρχουν από την πλευρά σας συγκεκριμένες ε, προτάσεις ή σενάρια που λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο σοβαρών κρίσεων στους κόλπους της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ ε, είναι έτοιμο να συμπεριλάβει και τέτοια σενάρια στις επιχειρήσεις σας ε, και αυτό ισχύει ε, και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Ευχαριστώ, κύριος Κέτλαμ. Ευχαριστώ πολύ. Με ικανοποίηση σημείωσα στρατηγέ ότι η ΕΠΑ δεν προτίθεται να ανταγωνιστεί το ΝΑΤΟ και υπάρχουν ορισμένα καλά παραδείγματα καλών ε, επιχειρήσεων ε, διαχείρισης κρίσεων. Όμως η αποφυγή του, της επικαλυψης το ΝΑΤΟ-ΕΠΑ ε, εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Οι πόροι, οι πιστώσεις προέρχονται από την ίδια πηγή, αν θέλετε, για τις επιχειρήσεις. Η ερώτησή μου αφορά τη δική σας εκτίμηση ε, των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Βιομηχανιών, γιατί η Επιτροπή συζήτησε διαμακρών την ανάγκη καλύτερου συντονισμού της παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ε, ενιαιοποίησης προτύπων, καλύτερο καταμερισμό εργασίας. Ποια είναι η γνώμη σας. Έχουμε επιτελέσει κάποια σημαντική πρόοδο εκεί. Ποια είναι τα προβλήματα κατά την κρίση σας. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη, τέλος, η αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν βλέπω πρόβλημα στην παράλληλη δομή το ΕΠΑ για λόγους διαχειριστικούς. Νομίζω ότι και οι δύο οργανισμοί έχουν κάποιες ελλείψεις και γι' αυτό είναι καλό να υπάρχουν παράλληλες προσεγγίσεις στην πολιτική αυτή. Κύριε Στρατηγέ, μια ερώτηση για την Αταλάντα, Αταλάντη. Νομίζω ότι ε, είναι ε, καλό αυτό που είπατε ότι είναι πολλοί στόλοι που δραστηριοποιούνται εκεί. Ε, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, θεωρείτε. Και ποιο είναι το επιχειρησιακό κόστος που πρέπει να υπολογίζομαι ώστε να συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε ε, Στρατηγέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Διαβουλεύσεις για μελλοντικές αποστολές. Ε, επανερχόμαστε στο ερώτημα το οποίο ε, έθεσε προηγουμένως ε, η κυρία Βουλευτίνα. Θα έπρεπε ειλικρινά να πω όχι διότι υπάρχει όπως ξέρετε ένα συνεχής διάλογος όχι σε δικό μου επίπεδο, στο επίπεδο Ξαβιέ Σολάνα και των υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά στην Επιτροπή σας παρακολουθείτε και ό,τι είναι ΠΕΣΚ ε, ούτως ή άλλως ε, είναι υπό τον έλεγχό σας. Στρατιωτικά εμείς κάνουμε προληπτική, προληπτικό προγραμματισμό και δεν έχουμε επαφές στρατιωτικές σήμερα για να καταρτήσουμε κάποια επιχείρηση. Απλώς είμαστε σε μόνιμη σχέση με τους ειδικού εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε όλες τις ζώνες κρίσεως. Τους συναντούμε, τους συναντώ και εγώ τακτικά και ο, στρατηγός Βίκη ο επικεφαλής του επιτελείου και κάθε φορά που έχουμε το, το αίσθημα ότι μπορεί να χρειαστεί να εμπλακούμε σε μία κρίση, ε, ξεκινάμε ε, προκαταρτικά και προληπτικά να ε, προγραμματίζουμε. Δεν υπάρχει κανένας τομέας αυτή τη στιγμή που να αποτελεί αυτή τη στιγμή ε, ένα κατεπήγον προγραμματισμού παρόλο που πέντε φορές τουλάχιστον προγραμματίσαμε ε, μήπως χρειαστεί να κάνουμε κάτι στην Παλαιστίνη, στην Μέση Ανατολή αλλά απεδείχθη ευτυχώς ότι, ήταν, ότι δεν υπήρχε λόγος σχετικά με, τους, ε, ε, με τον ε, πληθυσμό και τους πολιτικούς. Ξέρω ότι για τις δημόσιες προμήθειες γίνεται μία προσπάθεια να βελτιωθούν οι διαδικασίες μας. Η Γενική Γραμματεία προσπαθεί να καταρτήσει νέες διαδικασίες και στρατιωτικά είναι το πιο εύκολο γιατί υπάρχει συνεχής εξοπλισμός για να μπορούμε να τις αναπτύξουμε και δεν έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουν οι πολιτικοί. Ε, οικονομική κρίση και επικίνδυνο σενάριο στην Ευρώπη. Εδώ προσκρούομαι σε ένα νομικό βασικό θέμα το οποίο είναι το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και αμήνης διότι τώρα πολλά ναι. κράτη-μέλη θεωρούν ότι τουλάχιστον οι στρατιωτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο σε εξωτερικές επιχειρήσεις κρίσης και το αναφέρω σαν ένα αξιοπερίεργο διότι το σχέδιο της συνθήκης της Σαββόνας προβλέπει ε, ρήτρες αλληλοβοηθείας και ε, στηρίξεως πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα δηλαδή δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε ε, στρατιωτικές εμπλοκές ούτε καν για φυσικές καταστροφές προς όφελος κάποιου κράτους Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι απλούστατα διμερείς ε, επιχειρήσεις αλλά το ΝΑΤΟ έχει μία ευθύνη συλλογική αμήνης και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα για, μία, για έναν από τους συμμάχους εμπλέκεται το ΝΑΤΟ αμέσω. Άρα είναι φυσιολογικό το ΝΑΤΟ να προετοιμάζει παρόλο που ασχολείται πολύ περισσότερο με την εξωτερική προστασία της Ενώσεως από ότι ε, σε ε, κινδύνους όπως παραδείγματος χάρη είναι η τρομοκρατία. Για την τρομοκρατία υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και πολλά γίνονται μέσω διαδικασιών ε, στο επίπεδο του τρίτου πυλώνα. Υπάρχει πρόοδος αυτή τη στιγμή ο κύριος Βάης θα είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να σας ομιλήσει, διότι εγώ θα σας πω μόνο γενικολογίες και είναι ένας βασικός στόχος του γραφείου αλλά είναι πολύ δύσκολο να προοδεύσουμε και γι' αυτό εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω τι έχει να σας πει. Αν η ταλάντα θα συνεχιστεί, βεβαίως υπάρχει μία καταρχήν συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να συνεχιστεί ε, για ένα χρόνο 2009-2010. Ξέρουμε ακριβώς ε, ποια είναι τα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το 2010, διότι όλες οι χώρες μας έχουν ε, αναφέρει την συμβολή τους, άρα δεν ανησυχούμε για το πόσο θα οργανωθεί το θέμα αυτό και δεν κοστίζει και πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με τις σημαντικές οικονομίες της χώρες μας με, ε, περιορίζοντας τα λίτρα τα οποία πληρώνουν οι επιχειρήσεις και τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι ασφάλειες ε, είναι ένα κόστος το οποίο είναι πολύ ε, λογικό. Ευχαριστώ. Κύριε Στρατηγέ, όλοι εκτιμήσαμε τη σαφήνειά σας και ε, την ειλικρίνειά σας σε ένα βασικό θέμα. Σας συγχαίρουμε για την εργασία σας τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί δεν θα σας ξαναδούμε πριν αποχωρήσετε, αλλά σας συγχαίρω για την εργασία την οποία έχετε κάνει και ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Bien, nous allons passer à... Λοιπόν, τώρα προχωράμε σε ένα διαφορετικό θέμα το οποίο ε, έχουμε θίξει πολύ επιφανειακά αλλά θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε είναι ο κύριος Ιμπρέχ το υπεύθυνο του Κοινού Οργανισμού συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών διότι ο κύριος Μπελουάρ είναι σε μία συνεδρία στην έδρα του και θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό. Οπότε θα συζητήσουμε διάφορα προγράμματα εξοπλισμών που διαχειρίζεται η οργάνωσή σας, το α400M ή το Τίγρης, διότι στο παρελθόν η Επιτροπή μας ασχολήθηκε με τις στρατιωτικές μεταφορές ε, στον τομέα της αμήνης για να μπορούν να έχουν οι Ευρωπαίοι στρατιώτες το καλύτερο δυνατό πολεμικό υλικό και το ενδιαφέρον αυτή της παρουσιάσεώς σα είναι ότι θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε και μετά θα σας ρωτήσουν οι συνάδελφοι για διάφορα προγράμματα. Εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για τον Κώστε και τα προγράμματά του. Ε, όπως έχετε ήδη λάβει ε, ορισμένα υλικά, ίσως γνωρίζετε ότι ο ΚΑΡ σημαίνει Κοινό Οργανισμό Συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών είναι μία σύνμηση μία διεθνή, μιας διεθνής οργάνωσης που έχει σαν στόχο να διαχειρίζεται προγράμματα εξοπλισμών στον τομέα της αμήνης και της ασφαλείας ε, σε συνεργασία και ο Κώστε βασίζεται σε μία διεθνή συνθήκη και τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η ε, Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία. Έχει καταρτιστεί, είναι μια, ένα σχετικός νέος οργανισμός ο Κώστε και μπορούμε να μιλήσουμε για τις αρχές βάσει των οποίων ε, έχει δημιουργηθεί. Επισήμως ε, ιδρύθηκε το 1996 ε, μέσω διοικητικών διετάξεων και έχει ισότιμο καθεστώς από το 2001 οι αρχές ε, ε, είναι οι βασικές αρχές, δηλαδή αποτελεσματικότητα από πλευρά κόστους, εναρμονισμό στον τομέα των οπλισμών και ε, στην απέτηση των δυνάμεων και των τεχνολογιών για να υπάρχει απόδοση ε, και ε, μία διεθνής ε, ισοσκέληση και ο Κώστε είναι ανοιχτός και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα δε αυτό είναι στη διάθεση όλων. Οι αρχές αυτές ε, βασίζονται εις τη συνθήκη που κατήρτισε το κόστε και ε, περιλαμβάνονται ε, στην κάρτα μας που, είναι, που διέπει το σύστημα ποιότητάς μας. Υπάρχει σε τέσσερα σημεία Βόνη, Παρίσι, Τουλούζι και Ρώμη. Στη Βόνη είναι το κεντρικό μας γραφείο και ορισμένα προγράμματα, το Boxer, το Cobra, το Εσόρ και το Tigris. Στο Παρίσι βρίσκεται το Παρίσι Εσάφ και Φλέμ και στην Τουλούζη το A400M και στην Ρώμη ένα πρόγραμμα παρακολουθήσεως της Αφρικής. Κάθε πρόγραμμα λοιπόν είναι μία συνεργασία ε, μεταξύ τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές χώρες και επιπλέον υπάρχουν χώρες σαν την ε, συνεργασία για το α400μη ε, το, το, οποίο είναι και το πιο περίπλοκο πρόγραμμα. Έχουμε ένα διμερές πρόγραμμα το Boxer ε, γερμανο-ολλανδικό, η κόμπρα που είναι ένα γαλλικό, γερμανικό, αγγλικό και λίγο τουρκικό. Στο ΕΣΟΡ υπάρχουν ε, έξι χώρες που συμμετέχουν δεν θα σας το περιγράψω εκτενώς. Το α400M είναι ένα τεθωρακισμένο όχημα. Ε, το κόμπρα είναι ένα ραντάρ. Το ΕΣΟΡ είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού software defined radio για τους συγχρόνους ασυρμάτους και το Franco είναι γαλλοϊταλικό πρόγραμμα. Η ΕΣΑΦ είναι ε, μία ε, μία οικογένεια ε, των βλημάτων πυράβλων εδάφους αέρος και ε, το, ε, στο κόστε προσπαθούμε να καταλήξουμε στην καλύτερη επιλογή σε διάφορους τομείς και ε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, δηλαδή κάθε πρόγραμμα έχει το δικό του νομικό πλαίσιο και υπάρχουν ορισμένα, ορισμένες συμβάσεις που διέπονται από τη γαλλική, η αγγλική, η ιταλική νομοθεσία. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε ε, τις καλύτερες συνθήκες για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα. Υπάρχει μία ευέλικτη γεωμετρία τόσο στον τομέα του αριθμού των συμμετεχόντων, δηλαδή των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και όσο προχωρά το πρόγραμμα και εξελίσσεται. Προσπαθούμε να, ε, να προσαρμόσουμε τη μονάδα που το διαχειρίζεται και από πλευράς μεγέθους και από πλευράς υποστηρικτικών υπηρεσιών διότι χρειαζόμαστε λιγότερους τεχνικούς αλλά περισσότερους που γνωρίζουν πώς μπορούν να υπάρξει στήριξη των συστημάτων και διοικητική μέρισμα, logistics. Λοιπόν, ε, όλα αυτά τα θέματα προχωρούν καλά για τη διαχείριση των ευαισθητών πληροφοριών. Ε, είναι κάτι το οποίο ξέρουμε, διότι για το πρόγραμμα FREMT υπάρχει ε, μία, υπάρχουν φραγές και αν οι Ιταλοί δεν θέλουν οι Γάλλοι να δουν τι γίνεται τότε δεν μπορούν. Ε, προσπαθούμε δηλαδή να εφαρμόσουμε όλες τις ε, πληροφορίες ευαισθησίας και ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα και διαχειριζόμαστε διάφορους πόρους που έρχονται είτε από τα κράτη είτε από τον ιδιωτικό τομέα για να εφαρμόσουμε τα προγράμματα. Η θέση του Κώστε στην Ευρώπη είναι ότι προσπαθούμε να καταρτήσουμε πολλές διασυνδέσεις με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους και με κράτη με τα οποία προσπαθούμε να βρούμε μία διοικητική συμφωνία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου και συγχρόνως προσπαθούμε να καταρτήσουμε και μία συμφωνία ασφαλείας για τις ε, διαβαθμισμένες πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από πλευράς Συμβουλίου και ιδίως Επιτροπής. Έχουμε πολλές ε, σχέσεις ε, με την ΕΝΤΑ κατά τρόπον ώστε η έντα η οποία μελετά τις δυνατότητες εντοπισμού των κενών να μπορέσει να μας δώσει τις πληροφορίες στο κόστε ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην παρουσίαση ε, και στον καθορισμό με τον καλύτερο δυνατό ο τρόπο. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας, βασικούς μας στόχους. Καταλήγοντας λοιπόν, θεωρούμε ότι πρόκειται για μία ελαφρία ευρωπαϊκή οργάνωση όπου έχουμε συμφωνήσει ε, τα γενικά μας έξοδα να είναι κάτω του 1% και να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε όλες τις φάσεις και, και να υπάρχει ε, μία θαυμάσια εφαρμογή ε, της ε, corporate governance. Εάν λοιπόν δεν μπορέσω να σας απαντήσω σε ερωτήσεις που θα μου κάνετε, θα σας απαντήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Κυρία Λέζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι για το γεγονός ότι ήρθε να μας ενημερώσει ένας ειδικό. Είπατε ότι το κόστε ε, δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα και ως προς τις δαπάνες. Ε, αυτό ισχύει και για το φιλόδοξο πρόγραμμα του Airbus που μας κάνει να αμφιβάλλουμε αν είναι όντως αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Τώρα, συγκεκριμένη ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο σκέλος της προσφοράς για το Airbus. Ας πούμε, αν μειωθεί το ωφέλιμο φορτίο του Airbus αυτού, θα έχει νόημα πια το πρόγραμμα γιατί δεν θα μπορούν να μεταφέρονται, με τα γερμανικά τάγκς με αυτό, τα καθαρακισμένα πια. Δεύτερον, με αυτή την επιβράδυνση μήπως δημιουργηθεί μεγαλύτερο συνολικό κόστος και ποιο θα είναι αυτό, ποιος θα το επομιστεί. Και μετά την επιβράδυνση ε, ενδεχομένως ε, θα υπάρξουν ε, κάποια, κάποιες άλλες ε, στα πλαίσια του EDS ε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, περιορίζομαι σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις μόνο. Ευχαριστώ, κύριο Ζέμκε. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Εγώ είμαι Πολωνός. Η Πολωνία είναι από τις χώρες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το τι κάνει το κόστε. Ήδη συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα και το Υπουργείο μας ήδη εξετάζει και άλλα προγράμματα για ενδεχόμενη συμμετοχή. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Βλέποντας αυτά τα προγράμματα που κυρίως ενδιαφέρουν το κόστε, θα συμφωνήσουμε ότι τα προγράμματα έχουν, επιλογή, έχουν επιλεγεί καλά και τα βασικά προγράμματα αφορούν εξοπλισμούς προβληματικούς για όλους μας. Αυτό το βλέπουμε, φαίνεται σε όλες τις αποστολές. Το βασικό πρόβλημα τώρα, γνωστό σε όλους, πέρα από τις εθνικές φιλοδοξίες, είναι η χρηματοδότηση. Τα προγράμματα εξυγχρονισμού τρέχουν για αρκετά χρόνια και έχουν συσταθεί λίγα χρόνια πριν τότε τα δημοσιονομικά της Ευρώπης ήταν διαφορετικά. Και η οικονομική πραγματικότητα ήταν διαφορετική και σε επίπεδο κρατών μελών. Η ερώτησή μου είναι θεωρώ πολύ σημαντική. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη τώρα αντιμετωπίζουν μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα. Πώς μεταφράζονται αυτά στη χρηματοδότηση των ε, κυρίων προγραμμάτων σας, Box, Cobra, Airbus, Fregata το πρόγραμμα FREM, CONVERT. Μήπως θα επιβραδυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων <coughs> αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω αφορούσε την έθεση ήδη στην Έλφος και αφορούσε στο A400M και την τροποποίηση του προγράμματος και την αξιοπιστία του πρόγραμματος αυτού. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ στο ζήτημα των σχέσεων με την ΕΑΤΣ. Είναι πολύ σημαντική η σύναψη συμφωνίας ε, που έχει γίνει. Ε, διαρωτώ με λοιπόν κατά πόσο αυτές οι εξελίξεις υπό το φως των ε, νέων ε, διατάξεων που θα τεθούν σε ισχύ με τη Λισαβόνα για τις διαθρωμένες συνεργασίες ε, κλπ. δεν αφήνουν να προχωρήσουμε σε μια θεσμοθέτηση του Όκαρ Κώστε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την φυστάμενη φύση του που έχει κατά τον εξωτερικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ κύριε Βανμπάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε στην Ευρώπη για την ανάπτυξη νέου υλικού. Σίγουρα. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και με τις ΗΠΑ Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο εταίρος σε αυτό το τομέα. Ο Κώστε εδώ μπορεί να προαγάγει και τα διατλαντικά προγράμματα, ευρωαμερικανικά δηλαδή. Ευχαριστώ. Merci euh, Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σε ό,τι φορά την αποτελεσματικότητα θα πρέπει να δούμε την, ε, το κόστο κατά πόσο είναι αποτελεσματικό σε ό,τι φορά διαχείριση προγράμματος και αυτό το έχουμε καταδείξει. Όπως ε, το α400M, αν και υπάρχει τριετής καθυστέρηση και αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ε, τροποποίηση των συμβάσεων και των ε, ανταποδοτικών ωφελών στο... που αποτελεί και την βάση για τον διαχείριση προγράμματος. Τώρα για το κόστος, αν θα είναι πιο υψηλό ή όχι, ή για καθυστερήσεις περαιτέρω, προς το παρόν δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι οι συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν για μία περίοδο standstill, δηλαδή προσωρινής ε, διακοπής, όχι του προγράμματος αυτού καθεαυτού. Θα καταλήξουμε εξάλλου στην πρώτη δοκιμαστική πτήση στα τέλη του 2009, απλά έγινε μια ρίδα standstill αν θέλετε, μια διακοπή για το πρόγραμμα και υπάρχει εντολή για μια ομάδα που ονομάζεται JET της οποίας προεδρεύει ο στρατηγός ε, Λαμπαντουά είναι κάτι το οποίο έχει συστήσει το Βέλγιο για να προχωρήσει τις, ε, τις διαπραγματεύσεις και έτσι να έχουμε νέες ε, προϋποθέσεις ε, να υπάρχει μια αναδιάταξη αυτού του προγράμματος ε, για την μελλοντική διαχείριση. Τίποτα το ιδιαίτερα ευαίσθητο και απόλυτο δεν μπορώ να πω σχετικά με τις αυτές που ξεκίνησαν προχθές 1η Σεπτεμβρίου και ελπίζω να ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τις συμμετέχουσες χώρες που θα συνέλθουν τον Δεκέμβριο και να λάβουν την ε, τελική απόφαση. Οι εθνικοί διευθυντές ε, εξοπλισμών λοιπόν θα συνεδριάσουν και θα λάβουν την λόγο απόφαση. Να σας πω ότι ε, ο ΚΑΡ δεν λαμβάνει καμία απόφαση δρά εξ ονόματος ε, των κρατών ε, μελών τις αποφάσεις ε, τις λαμβάνουν οι, οι αρχικά ανώτεροι. Τώρα για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Όντως τα προγράμματα τροποποιούνται και σε αριθμό και σε υλικό και όλα αυτά φυσικά έχουν επιπτώσεις. Υπάρχει όμως μια συνεχής προσαρμογή. Τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν λαμβάνουν τις ε, αποφάσεις και δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιες είναι οι αποφάσεις που πρόκειται να λάβουν τα κράτη. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει επιβράδυνση των προγραμμάτων μετά από ε, οικονομικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένω να προκύπτουν. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Τα κράτη-μέλη πάντως στον προπολογισμό τους έχουν προβλέψει τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων και μπορεί σε κάποιο κράτος ε, να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί για να αλλάξουν ορισμένες παράμετροι και να έχουν ε, αντίκτυπο στο πρόγραμμα, αλλά σε ό,τι αφορά την ε, συνολική εξέλιξη του προγράμματος, αυτό συνεχίζει όπως ε, έχει προγραμματιστεί. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, σύντομα, οι φιλοδοξίες της ΟΚΑΡ αφορούν διάφορους τομείς. Ε, υπάρχουν έξι κράτη-μέλη Φυσικά θα μπορούσαμε να δεχτούμε στους κόλπους μας και περισσότερα μέλη. Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται από το Συμβούλιο, τον, το Εποπτικό Συμβούλιο. Τώρα την τελική απόφαση να περάσουμε από 6 σε 27 ή 28, δεν ξέρω εγώ πόσοι θα είμαστε όταν ε, ληφθεί η απόφαση. Την απόφαση αυτή έλεγα, την... Ε, θα τη λάβουν τα κράτη. Εάν τώρα οι χώρες που δεν ε, είναι μέλη του ΟΚΑΡ ζητήσουν να συμμετάσχουν, εντάξει αυτό είναι υποθετικό, μια υπόθεση κάνω, φυσικά και θα μελετήσουμε τα αιτήματά τους. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μελετήσουμε κάθε πρόταση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει δεν υπάρχει ακόμα κάποιο αίτημα συγκεκριμένο, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. κάτι τέτοιο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε, διότι τώρα έχουμε ιδιαίτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Εάν από 6 γίνουμε 27, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα λίγο μπλέκουν σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες Κοιτάξτε, στα προγράμματά μας συχνά συμμετέχουν αμερικανικές επιχειρήσεις. Τώρα διαχείριση ενός κοινού προγράμματος με τις ΕΠΑ δεν αποκλείεται διόλου. να έχουμε ως συμμετέχουσα χώρα την Μαλαισία ή την Νότια Αφρική, με καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θα έχουμε ως ε, εταίρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν το αποκλείει, θεωρητικά. Δεν θέλω να μπω τώρα στα πολιτικά χωράφια, αλλά μπορεί και να συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόγραμμα θα υπάρξει και ένας ε, Αμερικανός στρατηγός. Και σε όλες τις άλλες δομές θα εκπροσωπείται και η Αμερική, Μέση Πολιτή δηλαδή, και ο Να διευκρινίσω, Πρόεδρε, την φύση της απαντήσεώς μου, της ερωτήσεώς μου, που δεν ε, αφορούσε την ε, ένταξη και των 27 μελών στην ΟΚΑΡ αλλά μέσω ε, δομημένων ε, μηχανισμών θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί η ΟΚΑΡ ως έχει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην παραμένει εκτός που είπα, ε, στο εξωτερικό, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άποψη εξέφρασα. Oui, donc ναι αυτό μπορεί να πάει και πιο στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή είτε να υπάρξουν όλο και περισσότερα κράτη τα οποία θα συμμετάσχουν ή κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας ζητήσει να συγκεντρώσουμε όλες τις ενέργειες. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι στη βάση του κόστε τώρα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, άλλες επεμβάσεις σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση και για τις εξηγήσεις σας. Πρόκειται για σημαντικά θέματα επί των οποίων θα συζητήσουμε και με άλλους συναδέλφους σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατόπιν αυτού τη Δευτέρα στις 3 το απόγευμα θα συναντηθούμε με την Σουηδική Προεδρία και με την κυρία Σουηγινάρα.